Έκθεση Γκρέχ, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ χαίρομαι για το ότι ψηφίσαμε μια έκθεση για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τον καταναλωτή Σωστά στο σημείο 46 αναφέρεται πως το βασικό πρόβλημα είναι η πρόσβαση στο κεφάλαιο. Αυτό είναι σωστό γιατί εξακολουθεί να είναι το ένα hedge fund να βρει βεβαίως ε, πολλά εκατομμύρια από το να πάρει μια επιχείρηση ένα δάνειο 100.000. Οπότε θεωρώ πως ε, η έκθεση αυτή δεν ε, αποτελεί, δεν είναι μόνο λόγια, αλλά κινητοποιεί και την Κομισιόν να αναλάβει συγκεκριμένη δράση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φίγκερε εδώ κατόπιν. Προτίμησα το φαγητό, κύριε Φιγκερέιδο. Έκθεση Σμιτ τώρα. Ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένος πως ο διάλογος μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Για μένα σημαντικό είναι να μειωθεί ο αριθμός των νέων ανέργων, καθώς αυτό συχνά οδηγεί στο ότι δεν δημιουργούν οικογένεια ή καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια και αυτό βεβαίως επιτείνει και τις δημογραφικές τάσεις της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να προτιμούμε τους νέους ε, ανθρώπους ε, και να τους βοηθάμε να μπουν στην αγορά εργασίας. Επίσης η εκπαίδευση πρέπει να θεωρηθεί ως μέσο καταπολέμησης της ε, φτώχειας έτσι ώστε άνθρωποι να μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια τα οποία έχουν. Σας ευχαριστώ κύριε Μικολάσικ. Περνάμε λοιπόν σε μια επεξήγηση ψήφου για την έκθεση χάρμς. Δίνω τον λόγο στην κυρία, στον κύριο Κέλλη. Εγώ ψήφισα υπέρ, κύριε Πρόεδρε, για να κάνω το πράγμα το οποίο εγώ θεωρούσα σωστό. Όσον αφορά γενικά την πυρηνική ενέργεια θα έπρεπε να πω τα εξή. Οι πολίτε στη χώρα μου βρίσκονται σε σύγχυση σχεδόν. Όλοι είναι κατά τη πυρηνική ενέργεια ω αποτέλεσμα των καταστροφών στο Σέλαφιλτ και το Τσερνομπίλ. Γι' αυτό προτείνω στην Κομισιόν να ερευνήσει αυτό το ζήτημα, δηλαδή τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και να δημοσιεύσει ένα έγγραφο έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να αποφασίσουν ε, βασισμένοι στα γεγονότα και όχι στα συναισθήματα. Συμπερασματικά σας συγχαίρω για το εξαιρετικό σας έργο την πρώτη σας ε, ημέρα στην έδρα του Πρόεδρου. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη, ήταν πολύ ευγενικός να σας υπενθυμίσω πως κανονικά πρέπει να ζητήσετε επεξήγηση ψήφου πριν από τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ευρωπαϊκή κοινότητα θα βοηθήσει την ε, Λιθουανία, τη Σλοβακία και την Βουλγαρία σε σχέση με τις υποχρεώσεις του για την ε, θέση εκτός λειτουργίας των πυρηνικών ε, εργοστασίων όσον αφορά δε την Βουλγαρία. Βλέπουμε εδώ πέρα πως στόχος της πρότασης είναι να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια. Κύριε, κύριε συνάδελφε, οφείλω να, να σας αφαιρέσω το λόγο, γιατί εδώ πέρα αναφέρεστε σε τελείως διαφορετικό θέμα. Οπότε περνάμε τις επεξηγήσεις ε, ψήφου επί της έκθεσης ΝΓΟΚ. Ο κύριος Ταραμπέλα δεν είναι εδώ, οπότε τον λόγο έχει ο κύριος Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής ε, κατέθεσε πάρα πολλές τροπολογίες που ανέτρεπαν τελείως την έκθεσή του. Οτιδήποτε αφορούσε παραβιάσεις των ε, συνθήκων και επιτήρησης ε, των οικονομικών ε, αποκλήσεων ήθελε να τα σβήσει ο εισηγητής. Το όραμα του εισηγητή είναι να εξαντλήσει τελείως την οικονομία. Δεν θέλουν να αντιληφθούν 250 συνάδελφοι πως δεν υπάρχει αυτή η παραμυθένια χώρα που ονειρεύονται Έμα δάκρυα και υδρότα θα απαιτηθούν για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Και πράγματι δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στους ε, ψηφοφόρους μας. Πρέπει, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί το μακρύ χέρι που ανοίγει τις κάνλες του δημοσίου χρήματος. Ευτυχώς λοιπόν πήγε η ψηφοφορία όπως πήγε. Σας ευχαριστώ ο κύριος Γκίγκολ, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μιλήσει λίγο προηγουμένως, αλλά έχει φύγει. Κυρία Φόρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα είναι πολύ πιο βελτιωμένη η έκθεση τώρα για τα δημοσιονομικά από την αρχική διατύπωση. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα οικονομικά κίνητρα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους ελλείμματα. Αλλιώς ε, θα αντιμετωπίσουμε πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας, θα πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, δεν έχουμε πολλούς πόρους και όπου έχουμε θα πρέπει να τα δίνουμε σε τομείς όπου αποδίδουν όπως ε, έρευνα και ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα ενός γυράσκοντος πληθυσμού και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν ρυθίζουμε τα συνταξιοδοτικά. Θα πρέπει θέματα όπως η μετανάστευση ε, να αντιμετωπίζονται ευαίσθητα. Μπορεί να καλύπτει κάποια κενά στο εργατικό δυναμικό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, τα πραγματικά χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα σε τοπικό, τοπικό επίπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε την παγκοσμιοποιημένη ε, διάσταση του προβλήματος. Κλάις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση Χουάνγκιοκ και ο λόγος είναι νομίζω η ελαφρότητα εδώ πέρα με την οποία ζητάμε ακόμη περισσότερη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Πόσο πιο πολύ μπορεί να αποξενωθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους πολίτες όταν ζούμε τα προβλήματα της μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης. Πρέπει να γίνει μία ανάλυση κόστους-οφέλους για την μετανάστευση ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα, και τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα αρνούνται να υπολογίσουν αυτό το κόστος. Οπότε δεν υπάρχουν πλήρεις γνώσεις για αυτό το ζήτημα. Οπότε πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάμε και τα προβλήματα του τρίτου κόσμου από όπου φεύγουν οι εγκέφαλοι. Δηλαδή οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα ανέτησαν την κοινωνία έρχονται στην Ευρώπη. Πώς γίνεται να λυθούν αυτά τα πράγματα με ακόμη περισσότερη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ κύριε Κλάις. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Πεγιόντ. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ντότ. η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα εναντίον της έκθεση πρωτοβουλίας για την Ένωση για τη Μεσόγειο για πολλούς λόγους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια σταθερή Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Αλλά σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης, όταν η συγκυρία στην Ευρώπη είναι σε κατάσταση οικονομικής παραλυσίας, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσθετες δαπάνες οι οποίες συνδέονται με ένα τέτοιο σχέδιο. Οι μεγαλεπίβολες συναντήσεις των αρχηγών κρατών, οι γραμματείες, και τα πακέτα υποστήριξη δεν είναι ένα σχέδιο για αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εγώ υπέβαλα τροπολογία 5 ζητώντα η αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ με μια προτιμησιακή σχέση να μην προχωρήσει. Τη στιγμή που υπάρχει μια ανάγκη λεπτή ισορροπία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτόν τον τρόπο δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα να είναι αμερόληπτος μεσολαβητή η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διέλευση Παλαιστινίων Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφα. Ο κύριος Πόσελτ μετά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή των δεκαετίας του 80 ως νέος εισηγητής, ως νέος δημοσιογράφος είχα καλύψει το θέμα της απόρριψης της έτσι του Μαρόκου να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δούλευα τότε με τον κύριο Φων Χάψπουργκ που έλεγε ότι η Μεσόγειος πρέπει να είναι Μάρε nostrum και να ενώνει τις δύο όχθες της Μεσογείου. Σε μια βιογραφία του, του κυρίου Σαρκοζή έλεγε ότι είναι απαραίτητη η Ένωση για τη Μεσόγειο. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτήν την ε, λογική της σπατάλης όπως είπαν ορισμένοι. Θα πρέπει να δούμε ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι το σημαντικότερο εργαλείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε με σωστό τρόπο, θα πρέπει να την διαρθρώσουμε πολιτικά, όχι σαν μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Όπως ελέγχθη λοιπόν η, από τον Τζόρτζ είναι το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης η Μεσόγειος και επομένως πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση. Κύριε Λόφ, ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα την αρχική παράγραφο 12 στην έκθεση αυτή η οποία εκφράζει την ανησυχία της για την χρήση εθνικής κάθαρσης ως προήμιο για την αναγνώριση μαριονετών καθεστώτων στην Νότια Οσετία και στην Απχαζία. Η Ρωσία θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την κατάπαυση του πυρός πλήρως και να σταματήσει την πρόσβαση της ε, βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Απχασία και την Νότια Οσετία. Mm. Είναι απαράδεκτη και ταπεινωτική αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση προς τη Ρωσία να σεβαστεί την ακαιρεότητα της Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλαμ. Κλείνουμε λοιπόν τον κατάλογο των επεξηγήσεων ψήφων. Διακόπτω ως τις 3 ώρα το απόγευμα.